la Presidente. Allora, i lavori della... Ξεκινάμε λοιπόν το τελευταίο τμήμα των σημερινών εργασιών έκθεση Βάιλερ ε, για, την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Δίνω αμέσω το λόγο στην Μπάρμπαρα Βάιλερ για να κάνει την πρότασή της. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, και αξιότιμη Προεδρία. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα των σκιωδών εισηγητών της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ήτρε, Επίσης να ευχαριστήσω τους συνεργάτες και όλους που συνεργάστηκαν για αυτό το εξαιρετικό θα έλεγα αποτέλεσμα που πετύχαμε. Χωρίς την επικοδομητική και σωστή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Βελγική Προεδρία σίγουρα δεν θα καταλήγαμε σε αυτό το αποτέλεσμα όπως μπορείτε να φανταστείτε είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη ως εισηγήτρια με το αποτέλεσμα. Μια και φέρνει σημαντικές βελτιώσεις στην οδηγία και αφετέρου μια και νέες οδούς και πορείες ακολουθούμε για μια καλύτερη ηθική στις πληρωμές. Ο στόχος έχει επιτευχθεί θα έλεγα καλύτερα η τροχιά έχει χαραχθεί ώστε η φερεγγιότητα και η ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να βελτιωθεί των ΜΜΕ και να διασφαλιστούν οι επενδύσεις σε νέα προϊόντα, νέες θέσεις απασχόλησης και νέες διεργασίες. Τώρα γιατί ήταν αναγκαίο αυτή η οδηγία να βελτιωθεί. Ο νόμος του 2000 δεν ήταν δεσμευτικό, δεσμευτικός και ήταν λίγο αποτελεσματικός. Τα τελευταία χρόνια η ηθική πληρωμών σε σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη επιδεινώθηκε και μάλιστα πριν από την οικονομική χρηματοοικονομική κρίση η μεταρρύθμιση είχε, ήταν κάτι που το είχαν ευχηθεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στο πλαίσιο της Small Business Act εξέφρασαν επιθυμίες να διαμορφωθεί με πολύ καλύτερο τρόπο η ηθική πληρωμών στην Ευρώπη για τα αποτελέσματα. Αφενός πορευθήκαμε μια νέα πορεία. Έχουμε αυστηρούς κανόνες και κανονισμούς. Καταρχήν ισχύει η προθεσμία 30 ημερών με λίγες εξαιρέσεις και αυτές πρέπει να δικαιολογούνται. Έχουμε υψηλότερο ποσοστό επιτοκίου 8% για ληξιπρόθεσμες ε, οφειλές και έχουμε καταλήξει με μη γραφειοκρατικό τρόπο σε 40 ευρώ όριο. Και έχουμε πει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν με απλούστερο τρόπο να διεκδικήσουν και απαιτήχουν δικαίωση των δικαιωμάτων τους από ό,τι μέχρι τώρα. Η δεύτερη πλευρά είναι τα θετικά κίνητρα και τα νέα μέσα τα οποία πετύχαμε. Για παράδειγμα, όσοι είναι με καλή ηθική πληρωμόνα και να έχουμε και καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, εναλλακτικές ε, ε, δυνατότητες, δυνατότητα διαιτησίας είναι αυτό το νομοθέτημα μια συνεισφορά για better regulation, για καλύτερη νομοθεσία και ιδιαίτερα <clears throat> σίγουρα είναι κάτι το οποίο ικανοποιεί πολλούς. Σίγουρα υπήρχαν κάποιες ε, αντιπαραθέσεις και κάποια συγκρουσιακά θέματα. Να αναφέρω κάποια. Καταρχήν στο Κοινοβούλιο, στην αρχή, σίγουρα υπήρχαν μεγάλες διαφορές. Πολύ πάρα πολλές διαφορές απόψεων και οι 100 τροπολογίες από μόνες τους αποδεικνύουν το πώς έπρεπε να δοθεί αγώνας ε, για να επιληθούν τα προβλήματα. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν πάντα ικανοποιημένη με τη δική μας προσέγγιση για αυτά τα θέματα, αλλά νομίζω συνολικά καταφέρουμε να πετύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Προβληματικό όμως ήταν το Συμβούλιο από την άλλη πλευρά. Θα έλεγα ότι είναι θλιβερό ότι ότι είναι κρίμα ότι το Συμβούλιο το στόχο που είχε να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν, το πέτυχε, δεν τον πέτυχε, δεν τον πετύχαινε πάντα. Και ιδιαίτερα για τις μεγάλες πλούσιες καλά δομημένες χώρες όπως την Γερμανία και την Αυστρία για τις ενώσεις συλλόγους ε, ήταν επικοδομητικές ε, παρότι είναι αυτονόητο δεν μπορούσαμε πάντα να ακολουθήσουμε τις απόψεις και τις ε, προτάσεις τους. Επόμενα βήματα. Μετά την αυριανή ψηφοφορία αναμένουμε το Συμβούλιο να ε, να ευδοκιμήσει το θέμα στο Συμβούλιο με θετική ψηφοφορία και να ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη. Δεν αναμένουμε να περάσει η προθεσμία των δύο ετών για να τα υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη. Ήδη από τον Ιανουάριο 2011 πρέπει να αρχίσει η εθνική εφαρμογή όλων αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα λόγω στον Επίτροπο Ταγιάννη, ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση ολοκληρώνει μια σημαντική περίοδο εργασιών. Η Κομισιόν, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο αποφάσισαν από κοινού να δώσουν μια συγκεκριμένη απάντηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εφαρμόζοντας ένα τμήμα της πράξης που θα εγκριθεί αύριο το Small Enterprises Act υιοθετώντα δηλαδή μια οδηγία που θα επιτρέψει σε πάρα πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει τη Ευρώπη να αναπνεύσουν ανακουφιστικά. Ταυτόχρονα είχαμε μία άνοδο των απλήρωτων επιταγών, άνοδο κατά 8% πέρσι, 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Είχαμε απώλεια πιστώσεων, κάτι το οποίο βεβαίως θα έτσι μεγάλη δυσχέρεια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πολύ συχνά διατρέχουν τον κίνδυνο να τελειώσουν, να θέσουν τέλος στις δραστηριότητές τους επειδή ακριβώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους κυρίως εκ μέρου του δημοσίου ή των μεγάλων επιχειρήσεων. Νομίζω ότι τα θεσμικά όργανα θα δώσουν μια θετική απάντηση στην οικονομία της Ένωσης γιατί το να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη όταν θα υιοθετηθεί η προσέγγιση οδηγία θα διαθέσουμε γύρω στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι το οποίο νομίζω θα προωθήσει και την καινοτομία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως γνωρίζετε η πρόσβαση στις πιστώσεις αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας, οπότε θεωρώ ότι σήμερα το να υποστηρίξουμε την οδηγία, πρόταση οδηγίας της Κομισιόν αποτελεί μια σημαντική επιλογή για την οικονομία μας. Επειδή τελικά δίνουμε μια απάντηση και ελπίδα σε εκατομμύρια επιχειρηματίες και επιχειρήσεις στην Ευρώπη και εργαζόμενους βεβαίως οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σήμερα και αποτελούν την σπονδυλική στήλη τη οικονομία μα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Βελγική Προεδρία για την σημαντική τη συμβολή και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλου του βουλευτέ οι οποίοι σε αυτή την φάση συμμετείχαν ξεκινώντα από την κυρία Βέιλερ, τον κύριο Μπατασάρ, Ντε Άντζελης και όλου του κοιόδης εισηγητέ που επέτρεψαν να βρεθεί μια θετική λύση. Θεωρώ ότι χάρη στην εναρμόνιση των προθεσμιών πληρωμής του δημοσίου, δηλαδή η προθεσμία των 30 ημερών, θα δώσουμε μια πρόσθετη σημαντική ρευστότητα στις επιχειρήσεις. Αυτός ο κανόνας όμως θα πρέπει να οθήσει το δημόσιο που πληρώνει με καθυστερήσεις να υιοθετήσει άλλες καλύτερες μεθόδους διαχείρισης και ήδη προβλέπεται στον προπολογισμό μια αντίστοιχη γραμμή για αυτό το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν τακτικά να πληρώνουν τους ε, πιστωτές. Επίσης θεωρούμε ότι αυτές οι προθεσμίες θα επιφέρουν σε τελική ανάλυση και εξοικονομήσεις στις δημόσιε διοικήσεις. Ένα σημαντικό γεγονό είναι ότι το, οι ίδιες επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρώνουν τις δικές τους, ε, τα δικά τους τιμολόγια εντός 60 ημερών εκτός από συγκεκριμένε περιπτώσεις και για να ολοκληρώσω να υπενθυμίσω ότι οι χώρες μέλη είναι ελεύθερες να υιοθετήσουν τα πιο ευνοϊκά μέτρα προς τους πιστωτές ώστε να υιοθετηθεί οριστικά η οδηγία. Και θα πρέπει βεβαίως να υπάρχουν ή πιο σύντομε πρακτισμένε πληρωμών σε τελική ανάλυση ή σημαντικέ κυρώσει. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτέ, νομίζω ότι αυτή η οδηγία παρουσιάζει την βούληση της Ένωσης να δώσει μια σημαντική όθηση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να ξεπεράσουν μια οικονομική κρίση που η Κομισιόν προτίθεται να αντιμετωπίσει με μια σειρά παρεμβάσεων και μόλις ε, παρουσιάσαμε την ανακοίνωση για την καινοτομία. Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουμε και την ανακοίνωση για τη νέα βιομηχανική πολιτική γιατί δεν γίνεται να έχουμε καινοτομία και βιομηχανική πολιτική αν δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση στι πιστώσει. Και αύριο το Κοινοβούλιο, σε συμφωνία με την Προεδρία του Συμβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση σε αυτέ τι προσδοκίε. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπε. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Ντεάντζελη εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανικής Πολιτικής και Ενέργειας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Βάιλερ έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Με τις προτάσεις αυτές η Ευρώπη θέτει τέλος σε ένα μηχανισμό ο οποίος έχει γονατίσει τόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρεμβαίνει με στόχο την προστασία των μικρομεσαίων που είναι οι πιο θα έλεγα ευάλωτες στην ορμή της κρίσης, έχουν προβλήματα πρόσβαση στην πίστοση, έχουν προβλήματα ρευστότητας και οι καθυστερήσεις αποπληρωμής οδηγεί στο κλείσιμο πολλές επιχειρήσεις και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον τομέα της απασχόλησης μεταξύ των άλλων. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό αυτό που ε, καθορίζει το όριο σε 60 ημέρες ε, την υπερημερία με 8% και επιμέρους άλλες ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα κίνητρα, συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και καμία εξαίρεση. Αυτά είναι μέτρα για την υπεράσπιση των μικρομεσαίων, για την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού και θα πρέπει πλέον οι διάφορες χώρες να διασφαλίσουν την γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας αυτής που επιβεβαιεί τη χρησιμότητα της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπαλντασάρε για ένα λεπτό εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Ταγιάννη, κυρία Βάιλερ, συνάδελφοι. Είμαι υπερήφανος που συνεισέφερα και εγώ στην γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων σε αυτού του είδους την πρόταση οδηγίας που υποστηρίζει τις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις που καθορίζει σαφείς χρόνους αποπληρωμής που δημιουργεί κίνητρα αλλά και κυρώσεις σε αυτούς που καθυστερούν και αυτό ισχύει φυσικά και για τον ιδιωτικό τομέα και για τον δημόσιο τομέα. Αν όλοι οι εμπλεκόμενοι ε, πλήρωναν θα έλεγα άμεσα τα χρέη τους τότε θα είχαμε επιπλέον 300 δις ε, ευρώ στη διάθεσή μας. Λοιπόν, ε, δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να στρεβλώνουμε τον ανταγωνισμό όμως εφόσον δεν ισχύουν παντού οι ίδιοι κανόνες και αυτό είναι το νόημα της νέας οδηγίας. Να υποχρεώσουμε τις επιχειρήσεις και την δημόσια διοίκηση να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, να συνεισφέρουν στον αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισμού είναι μια μεγάλη επιτυχία η πρόταση αυτή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεπέρασε κάθε τύπου πιέσεις υπέρ των συμφερόντων των πολιτών και του ευρωπαϊκού παραγωγικού συστήματος. Ευχαριστώ. Ξεκινάει τώρα η συζήτηση με τους ομιλητές εξ των πολιτικών ομάδων να σας παρακαλέσω να σεβαστείτε το χρόνο σας γιατί έχουμε πάρα πολύ φορτισμένο, φορτωμένο συγγνώμη, πρόγραμμα και έτσι και αλλιώς στις 12 σταματάμε. Θα ξεκινήσουμε με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για δύο λεπτά Χάνσλικ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, τη συνάδελφη. Χαίρομαι που σήμερα έχουμε αυτή τη συζήτηση που ε, πρέπει να διεξαχθεί και έτσι έχουμε όλους όσους ενεπλάξαν σε αυτή την οδηγία και που γνωρίζουν ότι η συμφωνία δεν ήταν απλή υπόθεση και πολλές φορές τα προβλήματα ήταν γνωστά στα κόμματα, στις ομάδες για αύριο ελπίζω ότι θα έχουμε καλά μαντάτα για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μικρές επιχειρήσεις που θα έχουν την ευκαιρία να μπορούν να εισπράττουν τις οφειλές νωρίτερα και πιο έγκαιρα. Και έτσι σε κάθε κράτος μέλος θα είναι ίση η αντιμετώπιση. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι οι επιχειρήσεις βασίζονται σε μια κοινή ενιαία εσωτερική αγορά. Σε αυτήν δρούν. Και πολλές φορές ε, ε, ε, υπάρχουν διαφορές σε κράτη-μέλη. Θα πρέπει όμως οι επιχειρηματίες να έχουν την εγγύηση, να δίνονται τα εχέγγυα σε αυτές τις επιχειρήσεις, ότι έγκαιρα θα εξοφλούνται οι λογαριασμοί, άσχετα αν πρόκειται για Γερμανία, Γαλλία, Μάλτα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα ρωτήθηκα από έναν από τους δημοσιογράφους τι είναι εκείνο το οποίο αποτελεί τα κύρια μέσα το ενεργό στοιχείο αυτής, αυτού του νομοθετήματος που θα αλλάξει τα πράγματα στην αγορά. Αυτά τα δόντια, ας τα αποκαλέσω έτσι, αυτά τα μέσα είναι ότι η μέγιστη προθεσμία θα είναι 60 το μέγιστο ημέρες για την εξόφληση των γαρισμών. Είναι πολύ σημαντικό αυτά να μπορέσουν να λειτουργήσουν σε σχέση με τις επιχειρήσεις. Πρέπει οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν ότι έχουν απέτηση, θα έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν αποζημίωση σε περίπτωση που δεν θα θα τηρηθούν όλα αυτά και ότι ρήτρε ε, οι οποίε αποκλείουν σε κάποια σύμβαση την καταβολή αποζημίωση ή αποκλείουν ε, αυτή την προθεσμία δεν θα ισχύουν διότι θα πρόκειται για θέμητο ανταγωνισμό και καταχρηστικέ ρήτρε. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά αυτέ τι ρήτρε οι επιχειρήσει και μόνο έτσι θα μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά του. Η καθυστέρηση στι πληρωμέ πρέπει να είναι η απόλυτη εξαίρεση και όχι ο κανόνα. Αυτή η οδηγία θα δώσει το τώρα το σήμα θα σηματοδοτήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι έτσι θα βαίνουν καλώ. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ. Εξάματο ομάδα των Σοσιαλιστών, ο κ. Βερνό, για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον, την εισηγήτριά μας την κυρία Βέιλερ για την εργασία τη και για τον θαυμάσιο συμβασμό που βρέθηκε με το Συμβούλιο τη στιγμή που η αρχική πρόταση τη Κομισιόν παρουσίαζε σημαντικά σφάλματα. Θα ήθελα καταρχήν να μιλήσω για τρία σημεία σημαντικά τη οδηγία. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου για την ίση μεταχείριση ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Η Κομισιόν πρόβλεπε πιο βαριέ κυρώσει για τον δημόσιο τομέα τη στιγμή που θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια λογική κοινού Θα πρέπει να δούμε το θέμα από την οπτική των δημοσίων λογαριασμών και, του δημοσίου, και των εταιριών δημοσίου και της ανταγωνιστικότητας, ανταγωνιστικότητάς τους. Έχουμε την προθεσμία των 30 ημερών που παρουσιάζει σημαντικές περίπλοκες διαδικασίε πληρωμής για τις οποίες το δημόσιο δεν ήταν πάντοτε υπεύθυνο. Όσον αφορά τι προθεσμίες πληρωμών ήταν απαραίτητο να θεσπίσουμε την ρήτρα αυθαιρεσίας και το οποίο συμβαίνει συχνά όσον αφορά τις σχέσεις ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεγάλων επιχειρήσεων για τις ε, καθυστερήσεις πληρωμών το 8% και η αποζημίωση που καλύπτει τα έξω των μικρών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι κάτι το οποίο οθεί τις μικρομεσαίες να ζητήσουν αποζημίωση. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να μην σε θέση να το ζητήσουν αν δεν τρέχουν κάποιο κίνδυνο. Ελπίζω λοιπόν το κείμενο αυτό να αποτελέσει μια πραγματική πρόοδο όσον αφορά την βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μια σημαντική πρόοδο δηλαδή σε μια πιο αποτελεσματική νέα αγορά αλλά και πιο δίκαια. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ για την ομάδα των φιλελευθέρων Κρόιτσμαν, 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πίτρο Πεταγιάννη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αύριο θα ψηφίσει μια οδηγία για την καταπολέμηση καθυστερημένων πληρωμών που θα γράψει ιστορία πραγματικά. Είναι η πρώτη οδηγία που πολύ απλά με τρία λόγια, με τρεις προτάσεις μπορεί να εξεταστεί, να αναλυθεί. Πρώτον, στο μέλλον μέσα σε 30 ημέρες θα πρέπει να πληρώνει λογαριασμοί και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κάποια διαφορετική συμφωνία εκτός αν υπάρξει κάτι το οποίο θα απαιτεί ε, δικαιολογημένα μια μεγαλύτερη προθεσμία. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα συμβατικής ελευθερίας ε, προθεσμίες πάνω από 60 ημέρες ε, δεν θα επιτρέπονται πλέον εκτός αν αυτό έχει ρητά κατεξαίρεση συμφωνηθεί και όποιος μπορεί να είναι δυνατόν να εισπράξει αυτούς τους λογαριασμούς θα έχουμε τουλάχιστον σε περίπτωση μη τήρησης των ρητρών 40 ευρώ τα οποία θα εισπράττονται. Με αυτή την οδηγία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη βοηθούνται πάρα πολύ να βελτιώσουν τη ρευστότητά τους και να μην πρέπει να αναλαμβάνουν τόσες, τόσα δάνεια από τις ε, τράπεζες. Δεν θα είναι δυνατόν να επιβληθεί κάποια άλλη διάταξη σε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στα κράτη-μέλη σε σχέση με ανώτερες ε, προθεσμίες ε, δεν θα είναι δυνατόν να τηρήσουν ε, αποκλείς και μάλιστα λέμε ότι θα είναι δυνατόν η οδηγία όσον αφορά την καταπολέμηση των πληρωμών δεν είναι δυνατόν να δίνει την ευκαιρία να υπάρχουν και μεγαλύτερες προθεσμίες. Οι επιχειρηματίες που κάνουν δουλειές και συναλλάσσονται στην Ευρώπη ξέρουν, θα ξέρουν ότι μέσα σε 60 μέρες θα έχουν εξοφληθεί. Μεγάλη πρόοδο αυτή. Και αυτό ολοκληρώνει και την ενιαία εσωτερική αγορά μπορούμε να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, διότι βοηθούμε έτσι τι μικρομεσαίε επιχειρήσει με αυτή την οδηγία και την ενιαία εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματο της ομάδα των συντηρητικών, κ. Χάρμπορ, για δύο λεπτά. <clears throat> Πρόεδρε, από την ομάδα μου η μισή μου ομάδα και ο πρόεδρος της, ε, της Επιτροπής του Ανταγωνισμού συμμετείχαν σε αυτή τη δικασία και θέλω να ευχαριστώ την εισηγήτρια και τους συμμετέχοντες για αυτή τη θαυμάσια δουλειά. Θα ήθελα να περιλάβω εδώ και το Συμβούλιο και την Κομισιόν επειδή υπήρξε μεγάλη συζήτηση για τον κανονισμό αυτό. Νομίζω όμως ότι έχουμε να κάνουμε ένα κλασικό παράδειγμα εφιούς νομοθεσίας που αφορά την καρδιά του ζητήματος όσον αφορά δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει στα πλαίσια αυτή τη κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε ώστε οι χώρε μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία αυτή το ταχύτερο δυνατό. Δεύτερον, η Κομισιόν σωστά ανέλησε τα προβλήματα και τι επιτυχίε τη προηγούμενη οδηγία. Θα ήθελα όμω εδώ να παρατηρήσω κύριε και κύριοι ότι αυτή ήταν η πρώτη οδηγία όπου η συμφωνία των συστοσών της ε, Επιτροπής που καλούσε την Κομισιόν να παρουσιάσει την μελέτη επιπτώσεων είχε εισαγωστεί πλήρως και είχαμε αυτή την μελέτη επιπτώσεων η οποία σαφώς εντοπίζει εντόπιζε τους τομείς που θα έπρεπε να αλλάξουν και νομίζω ότι κυρίως η επιμονή αυτή τη στιγμή οι δημόσιες αρχές ιδιαίτερα θα πρέπει, θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές του, του ιδιωτικού τομέα και δεν μπορούν να καταχραστούν τις θέσεις τους σε σχέση με τους, προ, προμηθευτές αυτό είναι απόλυτα ουσιώδες και αυτό είναι η κύρια, το κύριο επίτευγμα θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Βελική Προεδρία και βλέπω ότι εκπροσωπούνται εδώ απόψε, επειδή απέκρουσαν αιτήματα από κάποιες χώρες μέλη συναδελφοί που προσπάθησαν να πετύχουν μια παρέκκληση από την προθεσμία των 60 ημερών και είπαμε στη Βελγική Προεδρία ότι δεν υπάρχει νόημα να έχουμε αυτή την οδηγία αν, δεν, αν το επιτρέψετε αυτό θα είναι κοινό νοήματο, αν επιτρέψει στι δημόσιε αρχέ να το κάνουν. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα καλό παράδειγμα ευφυού ε, νομοθεσία, συνάδελφοι, αλλά θα ήθελα να ολοκληρώσω κάνοντα δύο τελικέ παρατηρήσει. Πρώτον, θα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά αυτή η διαγεία και συνεκτικά σε όλε τι χώρε μέλη. Και δεύτερον, θα πρέπει να οδηγήσει σε μια αλλαγή νοοτροπία. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι πια αποδεκτό για τους μεγάλους πελάτες να εκμεταλλεύονται τις μικρές επιχειρήσεις με καθυστερημένες πληρωμές. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς θα πετύχει αυτή η οδηγία. Ευχαριστώ για την Ευρώπη των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας ο κύριος Ρώση για 1,5 λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Κιαγιάννη για τα επιχειρήματά του και τον ευχαριστώ. Πολλές φορές οι καθυστερήσεις προέρχονται όμως και από τη δημόσια διοίκηση και οδηγούν στην αποτυχία και στην πτώχευση επιτυχημένων κατά τα άλλα επιχειρήσεων με αλυσιδωτές δραματικές αντιδράσεις κοινωνικές κτλ. Πολλές φορές ε, στρέφονται δικαστικά εναντίον της δημόσιας διοίκησης η οποία τελικά είναι υπεύθυνη πολλές φορές για την αύξηση του κόστους και των τιμολογίων ιδιαίτερα στα πλαίσια της περίοδου κρίσεως και οικονομικής υφέσεως την οποία διανύουμε έχουμε αποτύχει να ελέγξουμε το θέμα των καθυστερήσεων, θα πρέπει να τιμωρούνται αυστηρά. Οι προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην πρόταση οδηγία βάζουν κάποια όρια, όχι άνω των 30 ημερών θέτουν τις 30 μέρες επίσης και τα, ε, για την προθεσμία για την πληρωμή των χρεών της δημόσιας διοίκησης προς τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης προβλέπουν συγκεκριμένες προθεσμίες και στον τομέα των μεταφορών της ενέργειας, των σχέσεων ανάμεσα, των συναλλαγών ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Θα πρέπει όμως τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την ε, οδηγία αυτή το ταχύτερο δυνατόν έτσι ώστε να οξυγονωθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πλέον γονατίσει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σετζέντι για τους μη εγγεγραμμένους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ουγγρική κοινωνία, ε, οικονομία έχει και αυτή πληγή από τις καθυστερήσεις εξοφλήσεων πληρωμών. Γι' αυτό χαιρετίζουμε αυτόν τον αυτή τη διάταξη που θα συνεισφέρει να βελτιωθεί η κατάσταση στην αγορά. Οι τροπολογίες και οι προτάσεις βελτιώνουν την, τον αρχικό στόχο, όμως κάποιες υπονομεύουν τις δυνάμεις εκείνες που πρέπει να διασφαλίζουν τον ρόλο των δημοσίων αρχών. Ιδιαίτερα σε αυτές τις αρχές δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να παρεκκλίνουν από την προθεσμία των 30 ημερών. Να μην υπάρχει μεγαλύτερη προθεσμία για αυτές. Όσον αφορά τις κυρώσεις, θα πρέπει να είναι ίδιες οι κυρώσεις για ιδιωτικές επιχειρήσεις και κρατικές δημόσιες επιχειρήσεις. Θα πρέπει έτσι να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διασφαλιστούν ότι θα εξοφλούνται για αυτούς τους λογαριασμούς. Και αυτό θα ήταν το καλύτερο αν θα ήταν δυνατόν να υπάρχει μια ε, δυνατότητα εξόφλησης ε, σε ε, σε, σε ενιαία προθεσμία. Υπάρχει όμως ε, πολλές φορές ε, ε, η επιβολή από κάποιους ισχυρότερους από μεγάλες επιχειρήσεις σε μικρές επιχειρήσεις επιβολή και 90 ημερών ακόμα και έτσι αυτά είναι καταστάσεις καταχρηστικές. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό θα έπρεπε σε οπωσδήποτε να ρυθμιστεί νομικά ότι όσον αφορά τις καθυστερήσεις ε, πληρωμών, όλες οι δαπάνες και τα κόστη που θα προκαλούνται θα πρέπει να αποζημιώνονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε τώρα τη συζήτηση με τους υπόλοιπους εγγεγραμμένους ομιλητές. ΣΒΑΜ για δύο λεπτά πρώτα. Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ήθιστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρχήν να ευχαριστούμε τους συναδέφους αλλά για αυτή την οδηγία πραγματικά πιστεύω ότι είναι θεμητό και δίκαιο να ξεκινήσουμε με αυτές τις ευχαριστίες. Πρώτα θέλω να ξεκινήσουμε με τις ευχαριστίες προς τον Επίτροπο Ταγιάννη. Σπάνια σε σχέση με το παρελθόν πολύ ανοιχτά και ειλικρινά λήφθησαν υπόψη οι επιθυμίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχεδιασμό των εργασιών τη. Ήταν αυτή η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπή κάτι το ιδιαίτερα χαρμό, χαρμόσυνο και καινοτόμο. Θέλουμε περισσότερε τέτοιε περιπτώσει καλή συνεργασία. Αλλά και εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεισφέραμε από την πλευρά μα, ώστε αυτή η οδηγία, όπω περιγράφηκε από αρκετού συναδέλφου, να μπορέσει να ευδοκιμήσει Μεταξύ τη Επιτροπή Ενιαία Εσωτερική Αγορά και Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ακολουθήσαμε μια κοινή στρατηγική, συνεργαστήκαμε στενά και επιτρέψτε μου να πω ότι η συνάδελφο Βάιλερ ω εισηγήτρια, ω εκπρόσωπο του ΕΛΚ, όχι μόνο ε, από πλευρά μου την χάνει των ευχαριστειών μου, αλλά και τη αναγνώριση ε, του έργου τη. Ε, και στο τέλο θα πρέπει για το έργο τη ω εισηγήτρια να πούμε ότι ήταν εξαιρετικό και εκπροσώπησε τα συμφέροντα του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν θα τα καταφέρναμε χωρί τη δική τη συνεισφορά σίγουρα. Ένα σημείο θέλω τέλο να επισημάνω. Έχουμε έναν τομέα που λίγο τον καλύψαμε. Είναι τα 40 ευρώ που σε καθυστέρηση συλλήβδην θα ισχύει και θα επιβάλλεται. Νομίζω ότι όταν θα φτάσει η ώρα εφαρμογή από πλευρά των κρατών μελών θα λάβουν υπόψη ε, οι καταναλωτές ε, αυτή τη δυνατότητα και θα πρέπει να επεξηγήσουμε σε αυτού τι γίνεται διότι τα 40 ευρώ σε κανονική α το πω έτσι ε, περίπτωση είναι κάτι το οποίο δεν θα εισπράττει. Θα καταβάλλεται μόνο όταν υπάρχει καθυστέρηση. Πρέπει να υπάρξει εδώ διαφώτιση του πληθυσμού των καταναλωτών να κατανοήσουν γιατί αυτό είναι προ όφελο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέλλη, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πολύ καλά σχόλια τα οποία έκανε νωρίτερα. Η πρόταση αυτή νομοθετική είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντική και θέλω να ευχαριστήσω την Μπάρμπαρα για τον τρόπο με τον οποίο έκανε την πρότασή της. Είναι υπόδειγμα σωστής και χρήσιμης νομοθετικής ρύθμισης. Θα βοηθήσει την οικονομία, θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα βοηθήσει ευρύτερα την κοινωνία και θα μας βοηθήσει να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας που τόσο λείπουν αυτή την εποχή είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τις αγορές να λειτουργήσουν πιο εύρυθμα, δεν θα ανεχόμεθα πλέον τις καθυστερημένες πληρωμές και θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να δουλέψουν καλύτερα και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Στη χώρα μου στην Ιρλανδία υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα πτωχεύσεων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα λόγω των καθυστερημένων πληρωμών. Αυτό συνέβη και σε μια εταιρεία με την οποία έχω κάποιες στενές σχέσεις και η οποία αναγκάστηκε να απολύσει πάρα πολλούς εργαζομένους εξαιτίας ακριβώς των καθυστερημένων πληρωμών για τις υπηρεσίες της. Να μην ξεχνάμε και τους γεωργούς. Έχουν και αυτοί υποφέρει από τις καθυστερημένες πληρωμές των ενδιαμέσων και των σούπερ Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να λειτουργήσουν θετικότερα ακόμα και στον τομέα των ε, τροφίμων. Ευχαριστώ πολύ. Κότσουσνικ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Πίτρο Πεταγιάννη, εγώ πιστεύω ότι εισαγωγικά θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εισηγητρία κυρία Μπάρμπαρα Βάιλερ για την πολύ θετική εργασία, εργασία της Νομίζω ότι με την τελική αυτή διαμόρφωση της πρότασης όλοι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Έναντι της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που φαινόταν ότι απήχε πολύ από την πραγματικότητα, καταφέραμε στη συνέχεια να προσαρμόσουμε αυτή την πρόταση στην πραγματικότητα. Καταφέραμε να αποσαφηνίσουμε και να διευκρινίσουμε με κατανοητό εύληπτο τρόπο το τι θα πρέπει να ισχύει και αυτό είναι ένα βήμα προς τα εμπρός. Και αν κάτι άλλο πρέπει να τονίσουμε είναι το γεγονός ότι έναντι της αρχικής πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταφέραμε την αρχή της ελευθερίας του, των συμβάσεων, της συμβατικής ελευθερίας να την διασφαλίσουμε. Και αυτό επειδή προβλέπεται ότι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αντιμετωπίζονται όπως και τα άλλα. Και αυτά τα όργανα θα πρέπει στο μέλλον έγκαιρα να εξοφρούν λογαριασμούς. Και αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα αποβαίνει προς όφελος των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Χαίρομαι ότι καταφέραμε να αφήσουμε στο πλάι, στο περιθώριο, κάποιες, ε, κάποιες διατάξεις που δεν ήταν σωστές και αναγκαίες ε, και ε, για την ίσπραξη ε, για παράδειγμα 5% επιπλέον σε περίπτωση καθυστερήσεων. Αυτό θα είχε οι επιβαντικές επιπτώσεις στους ήδη πιεσμένους πολύ προϋπολογισμούς. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν στην αναζήτηση ενός συμβιβασμού. Είναι σκόπιμο λοιπόν αυτό και χρήσιμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά ο λόγος του κύριο, στην κυρία Κορατσαπίλτ. Θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι, τους μετέχοντες στο Συμβούλιο, τον κύριο Ταγιάννη, Συμβουλίο για την Ευελιξία του και τους συναδέλφους για την επίτευξη αυτού του συνδυασμού στην πρώτη ανάγνωση, που είναι πολύ σημαντικό για μας, για όλους μας και τις επιχειρήσεις και εγώ ως επιχειρηματίας χαίρομαι γι' αυτό. Και γνωρίζω ως επιχειρηματία, επιχειρηματίες ότι η των πληρωμών είναι από τα κυριότερα εμπόδια των ε, επιχειρήσεων. Οδηγεί σε αβεβαιότητα και σε ζημιά στις επιχειρήσεις και αποτελεί μια μέγιστη επιτυχία το να περιορίσουμε τις πληρωμές της διοίκησης στις 60 μέρες επειδή απλά και μόνο έχουμε να κάνουμε ένα θέμα μείωση γραφειοκρατίας. Χαίρομαι επίσης επειδή οι μικρές επιχειρήσεις έχουν ένα πλαίσιο αναφοράς, επειδή πολλές φορές δεν μπορούσαν, δεν τολμούσαν να διεκδικήσουν τις πληρωμές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι βρήκαμε μια ισορροπία μεταξύ σεβασμού της ελευθερίας και ταυτόχρονα δώσαμε τα απαραίτητα εργαλεία στις μικρές επιχειρήσεις ώστε να μην κρατώνται όμοιρες από τις, όμοιροι, συγγνώμη, από τις, μεγαλύτερες επιχειρήσεις και να μην τις κυνηγούν για την πληρωμή των ε, οφειλών. Έχουν αυτή τη στιγμή λοιπόν το δικαίωμα να ασκήσουν αυτά που προβλέπονται από την οδηγία και να ζητήσουν αποζημιώσεις και κυρώσεις. Θα πρέπει λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Χάρμπορ, να έχουμε μια νοοτροπία εμπρόθεσμης πληρωμής, κάτι το οποίο θα επιτρέψει την καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και θα βοηθήσει όλους τους φορείς. Εμείς ε, στο Κοινοβούλιο χαίρομαι που λάβαμε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία πραγματικά θα κάνουν τη διαφορά που θα δημιουργήσουν απασχόληση και θα διευκολύνουν τις μικρομεσαίες. Τώρα Πρόεδρε, το σημαντικό ζήτημα τώρα είναι το Συμβούλιο και οι χώρες μέλη να αναλάβουν την ευθύνη τους και να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή στις χώρες τους των κανονισμών αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. πολύ. Η κυρία Ράπτη, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ξεκινάω με ευχαριστίες στην Μπάρμπαρα Βάιλερ, η οποία νομίζω ότι δίνει ένα χέρι βοήθειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ολόκληρης της Ευρώπης και άρα βοηθάει την ίδια την Ευρώπη σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για την οικονομία της ένωσης γίνεται μια πολύ σοβαρή και τεκμηριωμένη προσπάθεια να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. οι καθυστερήσεις πληρωμών ξέρουμε όλοι ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι αιτία να πτωχεύουν οι επιχειρήσεις αυτές και άρα να χάνονται θέσεις εργασίας. με μεγάλη δυσκολία αλλά ταυτόχρονα και με ακόμα μεγαλύτερη διάθεση συμβιβασμού προκειμένου να σωθούν θέσεις εργασίας καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία συμφωνία ίσως λίγο σκληρή αλλά σίγουρα αναγκαία και δίκαιη. αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι εγώ προσωπικά ως ελληνίδα έχω ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία για αυτό το θέμα. το γεγονός ότι η ελλάδα συμφώνησε σε περιθώρια πληρωμών που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν στενά εντό εισαγωγικών δείχνει τη μεγάλη δέσμευσή μας για την εξυγίανση της κατάστασης στη χώρα μου. ο γενικός κανόνας πληρωμών των 30 ημερών σημαίνει πάρα πολύ απλά πως πρέπει να αλλάξουν οι εσωτερικές μας διοικητικές διαδικασίες ελέγχου για την έγκριση των πληρωμών. η εξαίρεση των 60 ημερών ιδιαίτερα σε τομεί όπω η υγεία μα δίνει περαιτέρω το περιθώριο να χειριστούμε αλυσιδωτές διαδικασίες πληρωμών οι οποίες δεν ελέγχονται πάντα εύκολα. πιστεύω και θέλω να τα καταφέρουμε και αυτό γιατί το οφείλουμε στους εργαζόμενους και στους επιχειρηματίες της ελλάδας στους εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες της ευρώπης. πρέπει να δώσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις την ευκαιρία να δουλέψουν με περισσότερα κίνητρα και να δημιουργήσουν υγιή ανάπτυξη. ευχαριστώ. Καταρχήν, θα πρέπει αυτό σε σχέση με την εξόφληση των πληρωμών να το λάβουμε υπόψη για τους γεωργούς. Πρόβλημα αυτό, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρόκειται για την κατάσταση των γεωργών, για τις καθυστερημένες πληρωμές οι στόχοι, οι προθεσμίες είναι πολύ μεγάλες ε, και αυτό είναι ένα από τα αίτια. Γιατί η οικονομική κατάσταση πολλών γεωργικών επιχειρήσεων επιδεινώνεται. Οι γεωργοί δεν παίρνουν έγκαιρα τις εξοφλήσεις, τα χρήματα που τους χρωστάνε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έκθεση του κυρίου Μποβέ πρόσφατα ε, τοποθετήθηκε υπέρ των αγροτών, των γεωργών και είπε ότι δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 30 ημέρες η προθεσμία εξόφλησης. Θα πρέπει πραγματικά να μεριμνήσουμε να εφαρμόζεται αυτό στην πρακτική εφαρμογή καθημερινά, στη ζωή των κρατών μελών, διότι πρέπει να προστατευτούν οι γεωργοί από αθέμητες ε, πρακτικές, ε, από καταχρηστικές πρακτικές, ε, ιδιαίτερα από μεγάλες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν είναι εδώ ο κύριος Ζουβέν, ο κύριος Πυρίλο τότε για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε κύριε Επίτροπε Ταγιάννη, συνάδελφε Βέιλερ, η οδηγία για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις πυρομές, στις εμπορικές συναλλαγές αποτελεί μια σημαντική δράση και ισχυρή του Κοινοβουλίου μας το οποίο έγινε ερμηνευτής των ετοιμάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης που εδώ και χρόνια υποφέρουν αυτές τις καθυστερήσεις πληρωμών. Πολύ σοβαρό γεγονός το οποίο αποτρέπει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και οδηγεί σε αλυσιδωτή αποτυχία και πτώχευση επιχειρήσεων, επιχειρήσεις οι οποίες συνήθως είναι υγιείς και οι οποίες ήδη επιβαρύνονται από υψηλά επιτόκια από τις τράπεζες. Με τη συμφωνία Συμβουλίου, Κοινοβουλίου, οι επιχειρήσει θα μπορούν να βασίζονται τώρα σε κάποια σίγουρη προθεσμία όσον αφορά τι πληρωμέ. προθεσμίε οι οποίε θα πρέπει να τηρούνται και από τη δημόσια διοίκηση αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα. Η πρόταση οδηγία βεβαίω θα βελτιώσει την ε, ροή των επιχειρήσεων τα οποία θα μπορούσαν να επιχειρήσουν ευκολότερα στο ευρωπαϊκό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα ήταν λοιπόν σωστό να υπάρχει επίπτωση και αυτής της οδηγίας στις τιμέ καταναλωτή και εύχομαι τα ευρωπαϊκά όργανα και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα σε μια στιγμή κρίσης να βοηθήσει ακόμα περισσότερο επιτεχύνοντας τις προθεσμίες μεταφοράς της οδηγίας αυτής της εθνικής νομοθεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για ένα λεπτό ο λόγος στον κύριο Λάζακ. Σας ευχαριστώ, αξιότιμη Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Το αναγκαίο σχέδιο οδηγίας για το οποίο συζητούμε σήμερα είναι πολύ καλύτερο από το αρχικό σχέδιο. Καταφέραμε να πετύχουμε ένα συμβιβασμό για την αντιμετώπιση με ίδιο τρόπο των όσων θα αντιμετωπίζουν αυτές τις διατάξεις. Ενώ για τις επιχειρήσεις θα πρέπει να περιορίζονται σε 60 ημέρες αυτές οι προθεσμίες και μόνο κατ' εξαίρεση μπορούν να παρατείνονται, σε περίπτωση με συμβάσεις όσον αφορά δήμους και κοινότητες οι προθεσμίες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 30 ημέρες. Αυτό είναι λανθασμένο όμως πιστεύω εγώ, διότι όλοι θα έπρεπε να έχουν στη διάθεσή τους τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις το επιχείρημα ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, πιο ενεργοί, ε, διατάξεις με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για ε, να ωφελούνται από αυτές οι επιχειρήσεις δεν αληθεύει για τις περισσότερες πόλεις, μικρές πόλεις και δήμους και κοινότητες όχι μόνο στην Σεχία, αλλά και πανευρωπαϊκά. Το τελικό σχέδιο λοιπόν κατά κάποιο τρόπο ε, ασκεί διακριτική αρνητική μεταχείριση εις βάρος των μικρών πόλεων και δήμων και κοινοτήτων. Ευχαριστώ. Κόμι δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με την ανάγκη ενίσχυσης της οδηγίας 2035 για τη μείωση τουλάχιστον με σημαντικό τρόπο των προθεσμιών για την πληρωμή των εμπορικών συναλλαγών. Είναι προφανές σε όλους οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες των καθυστερήσεων πληρωμών στις εθνικές αγορές και ταυτόχρονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά έχουν λειτουργήσει αρνητικά στην αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα και έχουν θέσει σε αμφισβήτηση την ίδια τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας, δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σωστές όπως και αυτά που λέγαμε εμείς για να καταστεί το επιχειρηματικό κλίμα πιο κατάλληλο για την διεξαγωγή των ε, εμπορικών δραστηριοτήτων. Και επίσης θα πρέπει και ε, οι ρυθμίσεις, οι προτάσεις μάλλον για το 8% αυτό ε, επιπλέον σε περίπτωση καθυστερήσεων είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μερικά ερωτηματικά. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι οι προτάσεις αυτές είναι μια καλή ευκαιρία για κάποιες αλλαγές. Θα πρέπει η οδηγία αυτή να περάσει το ταχύτερο δυνατόν στην εσωτερική νομική αρχιτεκτονική των κρατών μελών και αυτό θα πρέπει να γίνει γρήγορα και με ομοιογενή τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Μπαστός δύο λεπτά. Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ καταρχάς την εισηγήτρια για την προσπάθεια την οποία έκανε. Θα ήθελα να συγχαρώ επίσης και όλους όσους πήραν μέρος στην επεξεργασία αυτής της συμφωνίας. Ήταν σαφές ότι έπρεπε μετά από δέκα χρόνια να τροποποιηθεί η προηγούμενη ενισχύη οδηγία και πρέπει να σταματήσουν ή τουλάχιστον να μειωθούν όσο περισσότερο γίνεται οι καθυστερήσεις στις πληρωμές. Τέτοιε καθυστερήσει είναι αδικαιολόγητε όταν εμπλέκονται κρατικέ επιχειρήσει. Οι αρνητικέ επιπτώσει είναι τεράστιε, είτε στο επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είτε στο επίπεδο τη εσωτερική ενιαία εσωτερική αγορά. Και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν τόσο περισσότερο, μια και βρισκόμαστε σε μια χρηματοοικονομική κρίση σαν αυτή που διανύουμε. Αυτή η νομοθετική λοιπόν δράση θα δώσει συνάφεια και νόμι, νόημα στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, στο σχέδιο Small Business Act. Θα βελτιώσει σίγουρα την ρευστότητα και φερεγγιότητα των επιχειρήσεων αυτή η οδηγία. Θα έχουν στα χέρια τους ένα αποτελεσματικό μέσα, μέσο για να διακρικήσουν τα δικαιώματά τους έναντι των κακοπληρωτών. Με αυτή την οδηγία η αρνητική πρακτική των ε, δημόσιων επιχειρήσεων θα είναι η εξαίρεση εκείνοι που είναι στις δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει στη διαχείριση να δίνουν το καλό παράδειγμα και πρέπει στους λογαριασμούς να, να εξοφλούν μέσα στην προβλεπόμενη διορία. Και έτσι λοιπόν σε σχέση με τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δώσουμε την δυνατότητα να εφαρμοστεί το δυνατόν ταχύτερα αυτή η οδηγία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ασάγε για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ επιχειρήσεις πραγματικά υφίστανται τα πάνδυνα από την καθυστερημένη πληρωμή και εξόφληση, ιδιαίτερα σε μια τέτοια κρίσιμη περίοδο. Αυτό θα έχει μεγάλες επιπτώσεις ε, στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω τις κρίσεις αυτές, αυτής μπορούν να χρεοκοπήσουν. Τώρα έχουμε την ε, πρόταση αυτή για την αντιμετώπιση των καθυστερημένων πληρωμών και σε σχέση με την διαφοροποίηση ε, ιδιωτικών επιχειρήσεων όσον αφορά τις και τις δημόσιες επιχειρήσεις. Υπάρχει και η προθεσμία των 30 ημερών και έτσι μπορούμε σε σχέση με μία ε, εξαίρεση που μπορεί να συμφωνηθεί μέχρι 60 ημέρες. Αυτή η δυνατότητα για μία μια παράταση εξόφλησης θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικό μέσο και το βλέπουμε αυτό στον δημόσιο τομέα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ε, καταλήξει στην κατάσταση που οδηγήθηκε η Ελλάδα, για παράδειγμα, που υπήρξε παράταση και μέχρι 165 ημέρες ε, για τέτοιες εξοφλήσεις. Ε, υπάρχουν βελτιώσεις όμως που έχουν συμμεθεί στην Ισπανία 150 ημέρες, στην Ιταλία 128 ημέρες και εταιρείε έπρεπε να, πλη, να πωλήσουν από τη, τα όσα είχαν ως περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουν να εισπράξουν ρευστά. Θα πρέπει να έχουν δικαιώματα όμως οι εταιρείε να μπορέσουν να ε, εισπράξουν αυτά τα χρεωστούμενα χωρίς να ε, προσφεύγουν σε μεσολαβητές και να προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για αυτές. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το βάρος αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί υπερβολικό για μικρές, μικρούς λογαριασμούς ε, και θα πρέπει να δούμε το δικαίωμα της ανάκτησης ε, όσον αφορά το πραγματικό κόστος ε, το οποίο ε, θα πρέπει να καλύπτεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι καλό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. διαδικασία Κατστιά υπάρχουν οκτώ εγγεγραμμένοι ομιλητέ. Αν σεβαστούν όλοι το ένα λεπτό, τότε θα μπορέσουμε να τους ακούσουμε όλους. Μπασέσκου. Στα πλαίσια της γενικότερης οικονομίας οι καθυστερήσεις έχουν λειτουργήσει αρνητικά για όλο το σύστημα αλλά και κυρίως για τις μικρομεσαίες. Ο στόχος λοιπόν είναι ευγενής θα έλεγα, φιλόδοξος και είναι οι κανόνες στα πλαίσια των εμπορικών συναλλαγών θα διευκολύνουν σαφώς ε, τη λειτουργία των επιχειρήσεων όπως επίσης και την ανάκτηση γενικά των ε, ποσών τα οποία χρωστούνται. Θα πρέπει βέβαια να μην υπάρξουν στρεβλώσεις και οι κανόνες να εφαρμοστούν σε όλους. Τα τελευταία χρόνια στη Ρουμανία έχουν ακριβώς λόγω αυτών των καθυστερήσεων κλείσει πάνω από 30.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καθυστερήσεις προέρχονται φυσικά και σε επίπεδο προϊόντων αγοραστέντων και υπηρεσιών και από πλευράς των κρατικών διοικήσεων. Και εκεί θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Ρόιτοβα, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Αύριο αυτή η οδηγία θα εγκριθεί και έτσι θα τεθεί τροχιά για ένα νέο πολιτισμό έγκαιρης εξόφλησης λογαριασμών και καταπολέμησης των καθυστερήσεων. Ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα το ε, εκτιμήσουν θετικά ότι έγκαιρα θα μπορούν ε, να εξοφλούνται και δεν θα πρέπει να περιμένουν ε, μήνες ολόκληρους για να πληρωθούν. Και έτσι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σε σχέση με το τέλος των 40 ευρώ και σε σχέση με την αποκατάσταση καθυστερημένων πληρωμών θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα πρέπει να ε, γίνει κάποιο λάθος θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι οι πληρωμές θα πρέπει έγκαιρα να ε, γίνονται. Χαίρομαι για το γεγονός ότι υπήρξε έγκριση του ε, γεγονότος ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ε, και οι δημόσιες επιχειρήσεις ε, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι η πιο σωστή αντιμετώπιση τους. Χαιρετίζω και συγχαίρω την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Τα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαιρετίζω και εγώ την έκθεση της κυρίας Βάιλερ, στην οποία εκείνο περί του οποίου πρόκειται είναι να δημιουργηθεί μια νέα ηθική και ένας νέος πολιτισμός όσον αφορά την εξόφληση λογαριασμών. Ας μην έχουμε όμως αυταπάτες. Είναι μεν ένα σημαντικό βήμα, αλλά όχι ικανό και ισχυρό, όχι επαρκές. Ξέρουμε ποιες δυσκολίες υπάρχουν. Είναι λοιπόν κάτι το πολύ σημαντικό αυτό το βήμα, αλλά δεν επαρκεί αφ' αυτού μόνο του. Είναι απόλυτα αναγκαίο να γίνονται έλεγχοι, να διεξάγονται έλεγχοι. Διότι είναι γνωστό ότι οι μικρές, μικρές επιχειρήσεις, για παράδειγμα στην Γεωργία, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες και βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση όσον αφορά την αλυσίδα αυτή και την αλυσίδα των τροφίμων και βρίσκονται στα χέρια ως όμοιροι των μεγάλων επιχειρήσεων. Όπως είπα, η έκθεση Βάιλερ είναι σημαντικό βήμα, αλλά είναι αναγκαίο να υπάρχει υποπτία και να υπάρχουν έλεγχοι. Ευχαριστώ. Άλβες για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα υπάρχουν σε πολλά κράτη-μέλη πολλές διαφορές όσον αφορά τους όρους πληρωμών στις επιχειρήσεις που ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Εμεί γνωρίζουμε ότι αυτή η κατάσταση δημιουργεί πολύ μεγάλες δυσκολίες για τις πληρωμές και έτσι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και πάρα πολλέ από αυτέ εκτίθενται σε πάρα πολύ μεγάλου κινδύνους. Είναι σαφέ ότι η σημερινή οδηγία που ήθελε να ρυθμίσει αυτό το θέμα και να περιορίσει ε, τα δεινά σημαίνει και σηματοδοτεί ένα βήμα προς τα εμπρός όσον αφορά την υλοποίηση των πληρωμών όχι μόνο μεταξύ των επιχειρήσεων και των σχέσεών τους με τις δημόσιες επιχειρήσεις αλλά επίσης και αυτό είναι θεμελιώδες σε σχέση με τις ε, σχέσεις των επιχειρήσεων μεταξύ τους. Έχουμε τώρα μια νομοθεσία που δίνει πρόσθετη αξία και προβλέπονται κυρώσεις για τις καθυστερήσεις πληρωμών. Και έτσι θα υπάρχει μια σημαντική ισορροπία που θα επιτευχθεί όσον αφορά εκείνους, εκείνες επιχειρήσεις που είχαν δεσπόζοντα ρόλο στις αγορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάσκα ένα λεπτό. Το νομικό περιβάλλον στις διάφορες χώρες μας διαφέρει και γι' αυτό ακριβώς και τα συστήματα πληρωμής και τα συστήματα ανάκτησης χρεών όλα αυτά είναι εντελώς διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά συνολικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποφέρουν. Στη δική μου χώρα υπάρχουν ε, δύο είδη δραστηριοτήτων που συστηματικά ε, σημειώνουν καθυστερήσεις. Καταρχάς ε, ο δημόσιος τομέας και δεύτερον υπάρχουν επίσης και ξένοι εργολάβοι ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα, που πάρα πολλές φορές φέρνουν τις ρωμανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση γιατί δεν έχουν αποθέματα για να πληρώσουν τους μισθούς των ε, εργατών τους, των εργαζομένων τους αν υπάρξουν κάποιες κάμψεις στην δραστηριότητά τους. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω να βελτιωθούν οι καταστάσεις αυτές. Ευχαριστώ. Κολίνο. Πρόεδρε, κύριε Ταγιάννη, συνάδελφοι, και οι Ιταλικές επιχειρήσεις και οι Ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις γενικότερα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα είναι οι επιχειρήσεις αυτές που έχουν μεγάλες ανάγκες σε ρευστότητα και δεν έχουν ιδιαίτερη πρόσβαση σε πίστοση τον τελευταίο καιρό και επηρεάζονται πάρα πολύ από τις κινήσεις αυτές, από τα χαρακτηριστικά αυτά της αγοράς δεν έχουν πολλά περιθώρια εναλλαγής δραστηριοτήτων και ακριβώς θα ωφεληθούν από τις προτινόμενες αλλαγές. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να βοηθήσουν τους πολίτες και τους επιχειρηματίες προς την ίδια κατεύθυνση. Οι δικαστικές ή, μάλλον οι διοικητικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες θα πρέπει να απλοποιηθούν και να δείχνουν γενικά οι κρατικές διοικήσεις σεβασμό σε αυτούς οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ή εργάζονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα πρέπει να μπορέσουν να παίξουν τον ρόλο που τους αναλογεί και στη σχέση συνεργασίας ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα θα ήθελα να δώσω στην κυρία Φλασίκοβα Μπένοβα. Όλοι όσοι έχουν εμπλακεί σε επιχειρηματικές δραστηριότητες γνωρίζουν τα πολλά προβλήματα τα οποία υπάρχουν από τις καθυστερημένες πληρωμές. Η κυρία Βάιλερ έχει κάνει πολύ σωστές προτάσεις τις οποίες υποστηρίζω και υποστηρίζω και τις τροπολογίες της. Καλό θα είναι να βρούμε όμως και περισσότερα μέτρα τα οποία να λειτουργήσουν θετικά, σαν θετικά κίνητρα. Σαν παράδειγμα, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να υποστηρίξουμε ε, και κάποιες ρήτρε ε, γρήγορων πληρωμών ή να ε, δημιουργήσουμε καταλόγους σαν παράδειγμα σωστών επιχειρηματιών που δεν καθυστερούν τις πληρωμές τους, σαν κίνητρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση. Γιάρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με την νέα ρυθμίση για την κατεαπολέμηση καθυστερημένων πληρωμών μπορούμε να πετύχουμε σημαντική βελτίωση για όλε τι επιχειρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώ για μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι αφόρητο να πρέπει να περιμένουν μήνε για την εξόφληση λογαριασμών. Χαίρομαι για το ότι έχουμε σταθερέ προθεσμίε πλέον και επιπλέον ε, κύρωση σε περίπτωση καθυστερημένων πληρωμών. Με αυτόν τον εναρμονισμό πανευρωπαϊκά συνεισφέρουμε πανευρωπαϊκά για την βελτίωση των ε, συναλλαγών που ιδιαίτερα θα ωφελήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε τα ερήφια, τους ε, εκείνους που παραβαίνουν ε, τις διατάξεις. Δηλαδή να δούμε ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν σκοπεύουν να συμμορφωθούν, αυτοί πρέπει λοιπόν να διωχθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η δικασία και πάλι ο λόγος στον Επίτροπο Ταγιάννη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση έστω και με διάφορες αποχρώσεις κατέδειξε την βούληση όλου του Κοινοβουλίου του Ευρωπαϊκού να υποστηρίξει αυτή τη νέα οδηγία που θα δώσει συγκεκριμένε απαντήσει στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Συγκεκριμένε απαντήσει εκατομμύρια πολιτών που θα επιθυμούσαν να προστατευθούν στην άσκηση του επαγγελματό τους από τα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα. Δεν μπορώ ως πρώην Ευρωβουλευτής παρά να χαρώ για την συνεισφορά όλων των Ευρωβουλευτών για την επίτευξη γρήγορου αποτελέσματος. σε συνεργασία με την Προεδρία. Να συγχαρώ όλους τους συμμετέχοντες βοηθού ευρωβουλευτών, γραφεία επιτρόπων, βελική προεδρία κτλ. Όμω δεν θα πρέπει να εφησυχάζουμε, όπω είπε κάποιο από του προαλήσαντε. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε ώστε αυτοί οι κανονισμοί να υιοθετηθούν το ταχύτερο δυνατό από τι χώρε μέλη. Το μέγιστο όριο είναι 24 μήνε. Ελπίζουμε να γίνει νωρίτερα και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Κομισιόν θα συνεχίζει να παρακολουθεί από κοντά τους τρόπους με τους οποίους θα μεταφερθεί η οδηγία και θα εφαρμοστεί. Και βεβαίως θα παρνεύουμε από αυτού στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συνεργασία προς την Κομισιόν και σας χαίρω για το θαυμάσιο αποτέλεσμα το οποίο επιτύχαμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ Επίτροπε. Ο λόγος στην εισηγήτρια, στην κυρία Βέιλερ. Αγαπητοί συνάδελφοι, για άλλη μια φορά ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι όλοι θα διαπιστώσουμε όταν αυτό το θέμα θα το έχουμε και θα το συζητήσουμε στις εκλογικές μας περιφέρειες, στις χώρες μας, αυτό το οποίο δεν είναι αυτονόητο για ευρωπαϊκά χαρτοφυλάκια θα συμβεί. Θα δοθεί πολύ μεγάλη υποστήριξη σε αυτή την πρόταση. Διότι οι καθυστερημένε πληρωμέ δεν είναι κάτι το, στο οποίο ασκούμε επικρίσει στι χώρε μα, αλλά είναι κάτι το αυτονόητο να πρέπει να μπορεί κάποιο να εξοφλεί λογαριασμού έγκαιρα. Άσχετα από ποιο τομέα γίνεται, για ποιο τομέα γίνεται λόγο και για ποια χώρα μιλάμε. Έχουμε μεγάλη λοιπόν συνένεση και συμφωνία επ' αυτού. Ευχαριστώ του συναδέλφου που ομόθυμα ε, ε, είπαν ότι συμφωνούν με αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι θετικό. Τρεις πτυχές θα ήθελα να αναφέρω. Όπως είπα στην αρχή της συζήτησης, αύριο θα θέσουμε την τροχιά τις ράγες προς αυτή, για αυτή την πορεία. Θα δούμε αν οι ελαφρύνσεις που εισάγουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για γεωργικές επιχειρήσεις για παράδειγμα και για χειροτεχνικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, αν αυτά επαρκούν για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους αυτές οι επιχειρήσεις. Θα δούμε και πώς θα λειτουργήσει η ελευθερία του συμβάλλεστε και των συμβατικών αυτών διατάξεων. Θα δούμε αν είναι κάτι το οποίο όλοι υποστηρίζουμε ή όχι. Θα δούμε και το 8% για καθυστερημένες πληρωμές αν επαρκεί ή όχι. Το Κοινοβούλιο ήθελε να επιβάλλεται 9%. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Ζητούμε να προσέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη-μέλη να μην μπορέσουν να αποδυναμώσουν και να νερώσουν εντός εισαγωγικών αυτή την οδηγία. Βλέπω να υπάρχει κάποια προοπτική επιτυχίας που διαγράφεται στον ορίζοντα. Άκουσα ότι η Ισπανία συντάσσει ένα νέο νομοθέτημα για αυτό το θέμα. Και ακούω ότι και από άλλα κράτη-μέλη το ίδιο συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, οπωσδήποτε στην κοινοβουλευτική μα επιτροπή θα έχουμε ένα monitoring, μια υποπτία, εποπτική δράση που θα ασκήσουμε, ελέγχου που θα ζητήσουμε να διεξαχθούν, ώστε να ξέρουν τα κράτη-μέλη μετά από αυτή την προθεσμία αν λειτουργούν τα πράγματα προ όφελο τη βελτιωμένη ηθική εξόφληση πληρωμών, ποιοι συμμορφώνονται και ποιοι όχι. Ευχαριστώ όλου που συμμετείχαν σε αυτό το θετικό Ευχαριστώ και την Βελγική Προεδρία και αυτό δεν αναφέρθηκε επαρκώ ίσω πιο πριν. Ξέρουμε πόσο επικοδομητικά και θετικά ε, διεξήγαγαν αυτές τις ε, ε, διαπραγματεύσεις. Μια μικρή χώρα το Βέλγιο, θα έλεγα όμω μια χώρα με ευφυεί μεθόδους και αποτελεσματικές μεθόδους για να επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έληξε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12.30.